και σε ό,τι αφορά τη συνδρομή στα κράτη-μέλη για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο επαφίεται στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Σέληξε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Βίκστρομ με θέμα το εφαρμοστείο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές Ρώμη 2. Το λόγο έχει η συγκήτρια, η κυρία Βίκστρομ, για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, Jag vill börja med att inleda och tacka min tidigare kollega Diana Wall. ευχαριστώ. Η συνάδελφος Βόλι εργαζόταν ε, για το θέμα αυτό μέχρι που έφυγε από το κοινοβούλιο. Πολύ ενδιαφέρον ε, ήταν για μένα να ε, μελετήσω όλη αυτή τη διαδικασία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την επικοδομητική του συνεργασία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να λύσουμε τα προβλήματα της Ένωση, Η συμβολή τους και τα σχόλιά τους και οι τροπολογίες τους τροφοδότησαν την έκθεσή μου και τώρα έχουμε μια λύση την οποία όλοι μπορούμε να υποστηρίξουμε και την οποία ε, ομόφωνα υπερψήφισε η Επιτροπή. Γιατί είναι τώρα όλα αυτά τόσο σημαντικά, ακριβώς επειδή οι διεθνείς περιπτώσεις ε, δυσφήμισης ε, είναι συχνό φαινόμενο στα κράτη-μέλη μας. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. Είδαμε ότι η Ευρώπη διαρκώς αυξάνεται, ο κόσμος κινείται ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ε, οι πολίτες μας έχουν οικογένεια σε άλλα κράτη-μέλη και νομίζω πως η δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης είναι κάτι το οποίο όλοι μας καλωσορίζουμε. Όμως... Αυτή την περίοδο περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να αναφέρουν και στοιχεία και γεγονότα που γίνονται σε άλλες χώρες. Ε, Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις διεθνούς δυσφήμισης και αριθμός ε, αυτών θα αυξηθεί στο μέλλον. Τώρα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο προκύπτει διαμάχη. Ποιες χώρα η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί. Εφόσον πρόκειται για διεθνείς νομικές υποθέσεις και θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο, θα πρέπει να υπάρξει ένα συμπλήρωμα στον υφιστάμενο, στον ισχύοντα κανονισμό Ρώμη 2. Και γι' αυτό το πράγμα συζητάμε σήμερα. Υπάρχει δυνατότητα της ε, επιλογής, δηλαδή ο κόσμος επιλέγει σε ποια χώρα θα δικαστεί ανάλογα με το ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό φυσικά και το βλέπουμε σε διάφορους τομείς να συμβαίνει. Ο κανονισμός Ρώμη 2 ε, συμφωνήθηκε το 2005 ε, και υπήρξε ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο. Δυστυχώς όμως δεν βρέθηκε λύση με το Συμβούλιο, το θέμα έμεινε σε κρεμότητα και πιστεύουμε πως πλέον είναι η ώρα για να δημιουργηθεί σαφήνεια ούτω, ώστε όλοι όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις να ξέρουν τι ισχύει. Η προβλεψιμότητα είναι ένας από τους βασικούς μου στόχους ε, στη δουλειά μου για αυτό το θέμα γιατί νομίζω πως αποτελεί την βάση για μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι ισχύει ε, και εμείς στην Επιτροπή μας ξεκινήσαμε με βάση τη θέση του Κοινοβουλίου το 2005 και προβήκαμε φυσικά σε παρέτητες ε, αλλαγές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν βασικοί κανόνες ξεκάθαροι, ούτως ώστε να ισχύει η να ισχύουν οι νόμοι της χώρας όπου ε, διαμένει ε, το συγκεκριμένο άτομο. Εάν είναι δύσκολο να καθοριστεί το ποια χώρα θα εκδικάσει την υπόθεση, τότε θα πρέπει ε, να υπάρχει δυνατότητα η δικαιοσύνη να ορίσει εκδότη των ΜΜΕ δεν μπορεί να, να, να περιμένουμε να γνωρίζει όλες τις νομοθεσίες όλων των κρατών. Ε, πρέπει όλοι να γνωρίζουν όμως ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και είναι σημαντικό να γίνονται σεβαστοί οι συγκεκριμένοι κανόνες. Θα πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματά μας και τις ελευθερίες μας. Η Κομισιόν νομίζω τώρα θα είναι σε θέση να δεχτεί ε, την πρότασή μας και ελπίζουμε ότι θα επανέλθει σύντομα με νέα πρόταση. Προσβλέπουμε σε αυτήν και μάλιστα περιμένουμε και πρόταση απόψε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βίξτρομ για την έκθεσή της ε, που τροποποιεί τον κανονισμό Ρώμη 2, που είναι και η βάση για το σημερινό ψήφισμα. Η συνάδελφός μου, η Vivian Redding, θα εξετάσει πολύ προσεκτικά τις συστάσεις σας. Στην έκθεσή σα προτείνετε τη συμπερίληψη μια διάταξη για τη σκοφαντική δυσφήμιση στην ε, Ρώμη 2. Ο κανονισμό Ρώμη 2 για το δίκαιο που ισχύει σε εξωσυμβατικέ ενοχές αποκλείει ε, την ε, σκοφαντική δυσφήμιση γιατί τότε δεν είχε καταστεί δυνατό μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου να βρεθεί συμβιβασμό στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη με το πόρισμα ότι πρέπει να υπάρξει ελάχιστη εναρμόνιση του ουσιαστικού δικαίου για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει μέγιστη σημασία στην εξασφάλιση του δικαιώματο έκφραση και ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα και τη προστασία τη ιδιωτική σφαίρα. Ο πλουραλισμό των μέσων μαζική ενημέρωση πρέπει να γίνει σεβαστό, όπω προβλέπει ο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όμω ταυτόχρονα το θεμελιώδε δικαίωμα τη ιδιωτική σφαίρα και αυτό είναι σεβαστό, γιατί προστατεύει από παραβίαση τη ιδιωτική σφαίρα ε, δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σωστή εξισορρόπηση αυτών των δικαιωμάτων. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν το ψήφισμά σα και θα το εξετάσουμε και θα το λάβουμε υπόψη όταν θα εκπονείουμε την έκθεσή μας για την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού ΡΟΜΗ 2 που θα εγκριθεί στα τέλη του 2013 προβλέπω. Ε, δεν βλέπω στην αίθουσα τη συνάδελφο κυρία Γκαλό και μεταβαίνω στου άλλους εγγεγραμμένου ομιλητέ, Το λόγο έχει ο κύριος ε, Ζεύκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι αλλαγέ τι οποίε προτείνει η κυρία Βίξτρομ στην έκθεσή τη, είναι πολύ σημαντικέ. Ε, για μένα τουλάχιστον ε, προσωπικά και αυτό για δύο λόγους. Ήμουν συντάκτη τη Έκθεση σε σχέση με τι Βρυξέλλε 1 και έχω πλήρη επίγνωση τη σημασία που έχει για την ασφάλεια δικαίου το να υπάρχουν ξεκάθαροι νόμοι για δεδομένη ε, αντιδικία, διαφορά. Ήμουν ε, επίσης δημοσιογράφος κατά το παρελθόν. Ε, έχω εργαστεί στην πολιτική τηλεόραση για μακρό χρονικό διάστημα και είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος και στην ελευθερία των μέσων μας και ενημέρωσης και στην ελευθερία της έκφρασης και του λόγου. Αλλά με ενδιαφέρει επίσης να είναι υπεύθυνη η δημοσιογραφία. Έχει υπευθυνότητα ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την επαρκή και αληθινή πληροφόρηση. Δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα μέχρι στιγμή ποιο δίκαιο πρέπει να είναι εφαρμοστέο για την περίπτωση κοφαντική δυσφήμιση. Σε μια εποχή όπου όλοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, όταν πολλέ πληροφορίε ε, μέσω του διαδικτύου ε, διακινούνται και δημοσιοποιούνται, φυσικά ε, μπορεί κανείς πολύ εύκολα να επιλέξει το εύκολο μονοπάτι αυτής ε, της διαδικασίας του forum shopping. Επιλογή δηλαδή. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εδώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα δικαιώματα των εναγόντων ή εναγωμένων. Υπάρχουν κάποια παραθυράκια αυτή τη στιγμή στη Ρώμη 2 και θα πρέπει να τα καταργήσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόσχεται ε, ότι του χρόνου ε, θα έχει προτείνει τις αλλαγές που εμείς επιθυμούμε. Ο είναι ο κύριος Ραφαέλε Μπαλτασάρε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Wickstrom για το έργο της, για την πολύ καλή έκθεση της και για, την, ε, για τους συμβιβασμού που πέτυχε. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να πληρώσει ένα κενό το οποίο δυστυχώ είναι πάρα πολύ εμφανές. Πρόκειται για τον κανονισμό ΡΟΜΗ 2. Το κενό λοιπόν αυτό προκύπτει σε ό,τι αφορά τις εξωσηματικές ενοχές και την εφαρμογή το συνειδητικό βίο και τα δικαιώματα του πολίτη. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο των προσωπικών δεδομένων. Μέσω του διαδικτύου μπορεί να ε, υπάρχει μεγάλη μετάδοση των προσωπικών στοιχείων. Αυτό έχει συνέπειες και για τη δικαιοσύνη και προκύπτει ε, θα πρέπει να προκύψει μια ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος έκφρασης και του προσωπικού δικαιώματος για τα προσωπικά δεδομένα. Καταλαβαίνω λοιπόν πόσο κατεπήγον είναι ο χαρακτήρα τη έκθεση. Υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει κατεπηγόντω να εφαρμοστεί ο κανονισμό Ρώμη 2. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, σε ό,τι αφορά ένα κέντρο για την επίλυση των διασυνοριακών τέτοιων προκλήσεων και προβλημάτων να μιλήσω για την εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται φυσικά κόστος, αλλά έτσι μπορεί κανείς ε, να προασπίζεται τα δικαιώματά του και να προασπίζεται και την ελευθερία τη έκφραση. Κυρία και Κούρια, για δύο λεπτά. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμεί οι Ιταλοί. Μα απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα αυτό, οπότε καταλαβαίνετε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο τη και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για αυτά που δήλωσε και για την αφορά που έκανε στην ε, σχετική ρήτρα. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η εισηγήτρια κατάφερε να βρει μια σωστή ισορροπία μεταξύ των προσωπικών ελευθεριών, της ε, ιδιωτικής σφαίρας και της νομικής βεβαιότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολύ συχνά βλέπουμε ότι υπάρχει ευρεστική παρανόχληση στο διαδίκτυο μέσω των νέων τεχνολογιών και αυτό παραβιάζει την ιδιωτική σφαίρα. Γι' αυτό λοιπόν η ιδέα του να μπορεί κανείς να το να μπορεί να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κέντρο για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδου ζητήματα είναι μια ιδέα πολύ ευπρόσδεκτη ασφαλώς. Πρόκειται λοιπόν για μια επιλογή υπέρ της ελευθερίας και υπέρ μία ε, ευνοϊκή λύση, οποία, η οποία μας βρίσκει σύμφωνους. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανυπομονούμε να σημειωθεί πρόοδο στο θέμα αυτό, καθώς ε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα εκκρεμή, τα οποία θα πρέπει να ζητούν. Ναι. Έχετε το λόγο, κυρία ευχαριστώ, Είναι πάρα πολύ καλό το ζήτημα αυτό της κυρίας Βίξτρομ. Προφανώ είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο στο οποίο να απευθύνεται κανείς για να βρει μία λύση, να ξέρει ποιος είναι υπεύθυνο, ποιος έχει δικαιοδοσία, ποια χώρα θα πρέπει να είναι αρμόδια για τέτοιες ενδεχόμενες ε, διαφορές και νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά η κυρία Βίκστρομ. Κρίμα που δεν ε, ζήτησαν το λόγο πιο πολύ συνάδελφοι. Φυσικά πρόκειται και ένα θέμα το οποίο είναι μία φυλακόμενο και ίσως να μην χρειάζεται να πάρουν πολύ το λόγο, αλλά νομίζω ότι αποτελεί προτεραιότητα το Κοινοβουλίο και χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ. κύριε. Σας παρακαλώ απαγορεύονται τα... οι επιφημίες, τα χειροκροτήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Ε, το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής ο Επίτροπος κ. Ντεγκούχτ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν ύψεστη σημασία και η συμμόρφωση επηρεάζει όλους τους ε, παράγοντες της Ένωσης και ιδίως τους πολίτες. Όλοι πιστεύουμε στην ελευθερία του λόγου, αλλά δεν πιστεύουμε ταυτόχρονα θα πρέπει να παραβιάσει τη ιδιωτική σφαίρα. Σημειώνει η Κομισιόν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβούμε στις απαραίτητε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους προτού ε, αναφέρουμε τον επόμενο χρόνο σε όλα αυτά τα θέματα. Σίγουρα θα είναι προτεραιότητά μα η ελευθερία έκφραση και η προστασία τη ιδιωτική σφαίρα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Βίξτρομ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, Επίτροπε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα και σύντομη αυτή συζήτηση στην Ολομέλεια. Πολύ δράμα προκλήθηκε με την έκθεση αυτή πέρσι την Άνοιξη, άρα περίμενα πιο έντονες συζητήσεις, αλλά στη τελική ανάλυση ομόφωνα πέρασε η έκθεση αυτή από την Επιτροπή. Ελπίζω παρόμοια να είναι και η υποστήριξη εδώ στην Ολομέλη αύριο. Όπως είπατε, θα πρέπει να πληρώσουμε ένα μεγάλο κενό. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης και αφετέρου να διασφαλίσουμε, να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα του ατόμου στην ιδιωτική σφαίρα, στα προσωπικά του δικαιώματα, στα προσωπικά του δεδομένα. Μίλησα με την Επίτροπο Βιάν Ρέντινγκ και ελπίζω σύντομα να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρειαστεί να κάνει πολλές προσπάθειες στο πλαίσιο αυτό, γιατί έχουμε ήδη υποβάλει μία πρόταση για το μέλλον. Ελπίζω να έλθει σύντομα αυτή η πρόταση, γιατί πραγματικά τη χρειάζονται οι πολίτες μας. Και στην ημέρα της Ευρώπης νομίζω ότι είναι σημαντικό να φροντίσουμε αυτό το νομικό κενό να πληρωθεί προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που μέτωσε τον λόγο και ανυπομονώ να δω τι θα γίνει αύριο στην ψηφοφορία. συνάδελφοι, η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30 το πρωί. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Ρινάλντι το, με θέμα το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής. Στην υπηρεσία της αλλαγής η εμπορική και επενδυτική